το θέμα, πέρα από πολιτικές ομάδες και κόμματα και ε, θα πρέπει να είμαστε εδώ πραγματικά ε, με πρόληψη και προφύλαξη και όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων να λύνουμε τα προβλήματα. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έλξε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εδώ. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή με θέμα η κρίση της ηφαιστειακής τέφρας. Περιμένουμε να καθίσει ο κύριος Επίτροπος για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη συζήτησή μας. Η συζήτηση θα ξεκινήσει με την συντάκτρια, την κυρία Τικάου. Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Κυρίε και κύριοι, ο κύριο Σίμψον ε, ζητεί συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν για τη συζήτηση αυτή για την κρίση από την ηφαιστειακή τέφρα διότι έπεσε θύμα των περιορισμών κυκλοφορίας λόγω των προβλημάτων στον χώρο του Νομένου Βασίλειου και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει να έρθει στο Στρασβούργο για τη συζήτηση αυτή. Θα μιλήσω λοιπόν εξ ονόματός του απόψε. Προφορική ερώτηση λοιπόν για την κρίση από την εφεστιακή τέφρα είναι πάρα πολύ επίκαιρη σήμερα, ιδίω ε, στο πλαίσιο τη συνεχιζό, της συνεχιζόμενης ταλαιπωρίας και προβλημάτων ε, στην ενέργεια κυκλοφορία, όπως και κατά την πρώτη έκρηξη του προηγούμενου μήνα του ηφαιστείου αυτού της Ισλανδίας, όπου είδαμε να κλείνει για έξι μέρες ο μεγαλύτερος ε, ναι, ο περισσότερο ενέργειος χώρο στην Ευρώπη. Τη επαύρη λοιπόν αυτή τη ε, αναστάτωσης βλέπουμε να ε, έχουμε συνεχιζόμενη παρατεταμένη ε, αναταραχή και αβεβαιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αεροπλοεία. Υπήρξαν μαθήματα τα οποία αντλήσαμε, διδάγματα τα οποία αντλήσαμε, αλλά η διάρκεια ε, και το κόστος ε, καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη, μια αναβαθμισμένη ανταπόκριση στη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εν ώψη και των επόμενων ε, μάλλον αναταραχών που θα υπάρξουν, επειδή δεν είναι διευκρινισμένη η διάρκεια, επειδή υπάρχουν προβλήματα και περιορισμοί για την ε, μετακίνηση των επιβατών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για την αντιμετώπιση ε, αυτών των συνεπειών είναι οι κατάλληλοι. Είδαμε κάποια ζητήματα τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο. Οι κανονισμοί για τους επιβάτες των αεροπορικών εταιριών προέβη ήταν ε, τελικά αποτελεσματική, διότι ε, αποτέλεσαν ένα δίκτυο ασφαλείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών των ε, ταραχών. Δεν θέλουμε να παραμένουν αποκλεισμένοι στα αεροδρόμια επιβάτε. Βέβαια, τέθησαν κάποια ζητήματα για το κατά πόσο οι αεροπορικέ εταιρείε πληρούν τι υποχρεώσει που έχουν απέναντι στου επιβάτε και τα δικαιώματα των επιβατών. Αποζημίωση, και θα πρέπει να δούμε τι ανατροφοδότηση λαμβάνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση των επιβατών και τι διασφαλίσεις μπορεί να παράσχει για το ότι πραγματικά τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την νομοθεσία οι αεροπορικές εταιρείε. Επιπλέον, η τρέχουσα κατάσταση εξέθεσε την ε, τροτότητα, αν θέλετε, της κατάστασης για επιβάτες οι οποίοι έχουν κλείσει σε τρίτες εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες και για τους οποίους δεν ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. Πώς προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το χάσμα αυτό στην νομοθεσία. Επίσης, πολύ νωρί, ε, σε πρώιμο στάδιο τη κρίση, αναγνωρίσαμε ότι υπήρξαν σημαντικέ οικονομικέ απώλειε, οι οποίε έπληξαν τι αεροπορικέ εταιρείε όταν έκλεισε ο εναέριο χώρο σε ό,τι αφορά πακέτο αποζημίωση για την αεροπλοεία, είναι ε, κάτι που με ανησυχεί γιατί θα πρέπει να δοθεί άμεσα η αποζημίωση αυτή στους θυγόμενου φόρεις και όχι απλά σε αεροπορικές εταιρείες. Και τα αντισταθμιστικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν ε, όλη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι κάποια κράτη ίσω ε, θούν πιο θετικά από κάποια άλλα το θέμα της χορήγησης οικονομικής βοήθειας σε αεροπορικές εταιρείες. Ποιες διασφαλίσεις μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις για να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στις αποζημιώσεις που θα δοθούν σε επίπεδο κρατών μελών και πώς θα εξασφαλιστεί το... Ε, πώς θα εξασφαλιστούν οι ισότιμοι κανόνες και η δίκαιη μεταχείριση. Επίσης, ποια διαδικασία θα πρέπει να τηρηθεί για ε, ζώνες απαγόρευσης πτήσεων Αυτές οι αναταραχές λοιπόν ακόμη και τα λεπορία ε, στις αεροπορικές μεταφορές ε, έχουν δείξει κάποιες αδυναμίες αυτών των διατάξεων για τη ρύθμιση και την, ε, τον καθορισμό ζωνών απαγόρευσης πτήσεων διότι υπήρξε υπερβολική προφύλαξη. Φαίνεται ότι μπορούν τα αεροπλάνα να πετάξουν ψηλότερα από ό,τι επιτρέπεται τώρα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια, τα τις τελευταίες εβδομάδες ε, έγινε σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι τόσο αυτή η διαφοροποιημένη προσέγγιση που βλέπουμε σήμερα. Επίσης γνωρίζουμε ότι ε, δίνει νέα έμφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συλλογή δεδομένων και στη μεθοδολογία ώστε να έχουμε μια πληρέστερη και αναλυτικότερη εικόνα αυτών των, ε, της διέλευσης των οπλάνων μέσα από την ηφαιστιακή τέφρα. Πρέπει επίση, επαναλαμβάνω, να γίνουν κάποια θέματα για τον ορισμό των ίδιων ζώνων απαγόρευση πτήση. Είδαμε επίση επίσης, τον μεγάλο συντονισμό που υπήρξε. Αναγνωρίσαμε επίση την ανάγκη μεγαλύτερη συνεργασία και σε άλλου τομεί, όπω παραδείγματο χάρη επιτάχυνση τη πρωτοβουλία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και για τη δημιουργία ενό ε, σχεδίου δράση κινητικότητα, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κρίση ε, σε αντίστοιχε περιπτώσει. Ο κύριος Κάλλας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πάρει το λόγο. Madam President, members. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σας κάνω μια επισκόπηση της εξέλιξης της κρίσης από το ηφαίστειο της Ισλανδίας και που έχει βέβαια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση επλήγει πολύ βαριά από τις ε, συνέπειες της έκρηξης του Ισλανδικού ηφαιστείου τον Απρίλιο που πλημμύρισε με φεστιακή τέφρα τον ε, αέριο χώρο της περισσότερης Ευρώπης ε, που έχει ε, αυτή η τέφρα σημαντικά έχει επιβλαβεί σωματίδια τα οποία επηρεάζουν τις κινητήρες των αεροσκαφών. Και γι' αυτό αναγκάστηκαν οι εθνικέ αρχέ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τι σχετικέ διαδικασίε, οι οποίε έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατέληξε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου όποτε αυτού που χρειαζόταν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα κινητοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει τα πλέον επίγοντα ζητήματα, λαμβάνοντα υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης και την ανάγκη για μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση με βάση το μοντέλο και τη διαδικασία για διαχείριση κινδυνών. Λάβαμε ε, στις 17-18 Απριλίου πρωτοβουλίες με τη συνεργασία της Eurocontrol και της Ισπανικής Προεδρίας για και προτείναμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Συνεπία όλη αυτή τη προσπάθεια, ε, με πλήρη συνεργασία με τα κρατημέλη και τον κλάδο, ορίστηκαν νέε διαδικασίε ε, σε μια έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Μεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι 19 Απριλίου του 2010. Αυτή η νέα διαδικασία εγκρίθηκε και έτσι ε, άνοιξε σταδιακά ο εναέριος χώρος με συντονισμένο τρόπο από τις 8 Απριλίου στις 20 Απριλίου του 2010. Μετά λοιπόν από την άμεση αυτή δράση εκπώνησε μια έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση ε, των επιπτώσεων ε, της κρίσης αυτής για την ε, αεροπλοεία. Έλαβε την πλήρη υποστήριξη του Συμβουλίου Υπουργών της 4ης Μαΐου. Η έκθεση αυτή εστιάζεται πιο πολύ στην αντιμετώπιση της τρέχουσα κρίση από την Πεστιακή τέφρα, ωστόσο προσπάθησε να αντιμετωπίσει ε, ταυτόχρονα και την ανάγκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αντιμετωπίζει αντίστοιχε κρίσει με αποτελεσματικό τρόπο και στο μέλλον. Αυτά που είδαμε τις τελευταίες δέκα ημέρες ε, δείχνουν ότι δεν έχει επιληθεί, ε, του αντίον μάλιστα η κατάσταση, γιατί το ηφαίστειο είναι ενεργό, εξακολουθεί να είναι ενεργό. Και το κλείσιμο ενέργειου χώρου συνεχίζεται, βλέπουμε, ανάλογα με τις καιρικέ συνθήκες που επηρεάζουν τη διασπορά του φεστιακού αυτού σύννεφου. Εμείς ε, παρακολουθούμε την κατάσταση. Υπάρχουν ε, τα συμπεράσματα της 4ης Μαΐου του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών και με τα χαράς να σας αναφέρω και κάποια πρώτα μέτρα τα οποία λάβαμε. Υπάρχει μονάδα συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία από την 11 Μαΐου καταλήγει σε κάποιες τελικές διευθετήσεις, τις οποίες θα τις καθορίσουμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε τα λεγόμενα λειτουργικά τμήματα, ένα αεροχώρο τα οποία η Επιτροπή Ενίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ε, Ουρανού τα ενέκρινε. Υπάρχει επίσης και μία άλλη ομάδα ε, που συστάθηκε στις 7 Μαΐου Έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπλοείας που θα καθορίσει δεσμευτικά πρότυπα και μέτρα ε, για τις ε, οριακές τιμές σε ό,τι αφορά την εφεστιακή τέφα. Θα πρέπει να δούμε τώρα πώς τα διάφορα μοντέλα ε, πρόβλεψης και διασποράς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις επειδή υπάρχουν και άλλα που πρέπει να δούμε, θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των ε, συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών και θα έχουμε και ακόμη και άλλα μέτρα τα οποία θα επεξεργαστούμε. Τώρα το λόγο θα πάρουν ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ξεκινώντας ο κύριος Μαρινέσκου για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκρηξη ηφαιστειακή του Απριλίου μας έδειξε ότι οι αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένες για μια σωστή απάντηση σε μια τέτοια κρίση. Δεν υπήρξε ευελιξία στην αναπροσαρμογή των ε, πτήσεων. Η, η υιοθέτηση των μέτρων έγινε παρά την αντίρρηση των ε, κρατών ε, μελών. Ε, και όταν προέκυψε η κρίση φάνηκε η ανεπάρκεια αυτών των μέτρων. Και όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, χρειαζόμαστε αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των αεροπορικών μεταφορών που να μην λαμβάνει υπόψη ε, τα εθνικά σύνορα. Αλλά ε, προς το παρόν δεν είναι αυτό το πρόβλημα, η ταχεία εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν εδώ μεταξύ ε, μπορεί να είναι πολύ θετικά. Ε, πρώτα απ' όλα η δημιουργία λειτουργικών τμήματων του εναρίου χώρου που να ε, τηρήσουν την προθεσμία μέχρι το τέλος δηλαδή του 2012. Χρειαζόμαστε όμως και τον οδηγό που προβλέπει ο κανονισμός. Και δυστυχώς ε, η απόφαση της 4ης Μαΐου δεν αναφέρεται σε αυτόν τον οδηγό. Η απουσία αυτών των κατευθύνων γραμμών μπορεί να είναι ε, ο λόγος που επικαλούνται τα κράτη-μέλη για τις ε, μεγάλες καθυστερήσεις που ε, υπάρχουν. Επιπλέον όμως όλων αυτών χρειάζεται ένας έλεγχος της ε, ενέργειας κυκλοφορίας ε, μεταξύ ε, και συντονισμός μεταξύ γειτονικών λειτουργικών θυμάτων του εναρίου χώρου χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις. πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο προς το παρόν να προβλεφθεί ένας ε, τρίτος κανονισμός που να ενώνει όλα αυτά τα τμήματα. Μια τέτοια προσέγγιση ε, ε, θα επιτρέψει επίσης η εφαρμογή αυτού του συστήματος να γίνει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με το μικρότερο κόστος. Τα τελευταία κράτη-μέλη θα προσχωρήσουν φυσικά και αυτά στον χώρο Σέγγεν από την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απάντησή σας καταρχάς κύριε Κάλας. Βέβαια δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ζητήματα αρκετά και θα ήθελα να επαναλάβω κάτι. Απουσιάζει ο συνάδελφος Brian ε, Simpson και αυτό δείχνει ότι το θέμα παραμένει επίκαιρο. Ότι ε, είναι απρόβλεπτες ε, οι συνέπειες της κρίσης της υφησιακής τέφρας και του νέφους και είναι απρόβλεπτες συνέπειες για τους πολίτες και για την οικονομία μας και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα το καλοκαίρι. Να κλείνει ένα αέριος χώρος ε, εν μέσω των διακοπών. Και θα πρέπει να βρούμε διαρθρωτικά μέτρα που να βοηθούν την εναέρια κυκλοφορία και γενικότερα το σύστημα των μεταφορών και να το κάνουν πιο αποτελεσματικό. Θα επανέλθω σε αυτό. Ε, θα πρέπει όμως επίσης να ε, έχουμε καλύτερη διαχείριση της κρίσης. Το είπατε προηγουμένως αυτό, ότι θα συστηθεί ένα τέτοιο γραφείο ή μονάδα συντονισμού, την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε περισσότερα. Μπορείτε λίγο να μας πείτε Ποια θα είναι η εντολή που θα τους δώσετε, ποια θα είναι τα πρώτα καθήκοντα αυτής της υπηρεσίας. Τα γεγονότα του Απριλίου έδειξαν ότι ο συντονισμός μεταξύ των ενεχομένων πλευρών, αεροδρόμια, εταιρείε, ταξιδιωτικές, ταξιδιωτικά γραφεία δεν είναι δεδομένος, πάει στραβά, δεν υπάρχει μηχανισμός ε, για να ενημερώνει τι πρέπει να κάνει κάποιος και οι άνθρωποι που έχουν αποκλειστεί ε, σε αεροδρόμια δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους. Χρειάζεται λοιπόν καλή ε, προσπάθεια για να λαμβάνονται γρήγορα οι σωστές αποφάσεις και να γίνονται οι σωστές επαφές. Το ίδιο ισχύει και για τον επαναπατρισμό ε, ταξιδιωτών. Δεκάδες χιλιάδες είναι αυτοί. Κάπως πρέπει να έχουμε ένα σύστημα να τους διευκολύνουμε. Τα δικαιώματα των επιβατών επίσης πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχει μεγάλη ρύθμιση η νομοθεσία Ευρώπη και αυτό είναι θετικό, αλλά υπάρχουν ακόμα κενά και παραθυράκια Συζητήσαμε για τι τρίτε χώρε για εταιρείε που εδρεύουν σε τρίτες χώρε και δεν ε, διέπονται από τη δική μα νομοθεσία. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα δικαιώματα των επιβατών να τα εντάσσουμε και στι συμφωνίε τι αεροπορικέ με τρίτε χώρε. και κάπω να ε, εφαρμόζεται και στα κράτη-μέλη η νομοθεσία, έτσι. Αυτή τη βδομάδα μάθαμε ότι οι Ιταλικέ αρχέ έβαλαν πρόστιμο στη Ράια Νέα. Εντάξει, καλά νέα είναι, αλλά τα άλλα κράτη-μέλη τι κάνουνε. Μπορείτε να μας δώσετε μια αξιολόγηση. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά διαρθωτικά μέτρα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Ο ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό που φτιάχνεται αυτό το καιρό, αλλά μην ξεχνάμε και το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομο δεν ε, αποδείχθηκε εναλλακτική λύση και αυτό οφείλεται σε πολλά πράγματα. Είναι διαφορετικά τα συστήματα, ε, τεχνικά και άλλα. Εντάξει, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Επίτροπε, αυτό και έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μα αλλά θα ε, σας υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλντράουι. Τώρα έχει το λόγο για την ομάδα των φιλελευθέρων ο κύριος Μέσνερ. Η κυρία, η κυρία Μέσνερ, με συγχωρείτε, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μετά την έκρηξη ε, του ηφαιστείου το συζητήσαμε αμέσω το θέμα αυτό μαζί σας και τα προβλήματα. Και είδαμε διάφορα προβλήματα με την κρίση. Είδαμε ας πούμε ότι πόσο σημαντική είναι για τις μεταφορές η αεροπορία. Διότι ε, δεν ε, αποκλείστηκαν μόνο επιβάτες αλλά και ανταλλακτικά εμπορεύματα. Η BMW στη Γερμανία έχει πρόβλημα γιατί δεν μπόρεσε να στείλει τα ανταλλακτικά της. Δηλαδή χρειαζόμαστε όλα τα μέσα μεταφοράς και το αεροπλάνο για όλη την οικονομική ζωή. Επιπλέον μέρε ολόκληρε ε, να μην πετάνε τα αεροπλάνα, πέντε μέρε οι, οι, οι εταιρείε μπορούν να, το ανεχτούν, αλλά αν ήταν 20 αυτές τις μέρες θα είχε καταρρεύσει όλο το σύστημα, όλες οι εταιρείε για μεγάλο διάστημα. Τώρα προς το παρόν δεν μιλάμε για αποζημιώσεις, ε, λέμε θα το επομιστούν το κόστος οι εταιρείε. Τα δικαιώματα των επιβατών τα είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ε, τώρα αυτοί έζησαν στο πετσί τους τι σημαίνει αυτό. Ε, σε έκτακτες περιστάσεις, ε, αν έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει για τους επιβάτες, για τις αποζημιώσεις, για τις εναλλακτικέ λύσεις, για τις αντισταθμίσεις κτλ. όπως τα είχαμε αποφασίσει. Τώρα όμως θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, ο ευρωπαϊκό ουρανό. Ε, δεν έχουμε ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, ένα αέριο χώρο και αυτό ε, πραγματικά μας πόνεσε και ήταν ε, οδυνηρή αυτή η απώλεια. Βέβαια δεν μπορούμε ε, αν είχαμε ε, ενιαίο ουρανό, δεν θα σημαίνει ότι δεν θα ε, είχαμε την έκρηξη του ηφαιστείου, αλλά θα έχουμε καλύτερο συντονισμό. Εντάξει, ε, τώρα έχουμε να συντονιστεί, είπατε, και αρχίζει να εργάζεται η υπηρεσία αυτή και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ενιαίο εναέριο ουρανό. Εσείς ε, πώς το εκτιμάτε αυτό χρονικά, μέχρι πότε θα χρειαστεί. Βέβαια μπορείτε να μου δώσετε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά μήπως τώρα και πάλι ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να βοηθηθεί και με καλύτερο συντονισμό που ζητάμε τόσο καιρό στην Ευρώπη και το έχουμε στα χαρτιά να συμβάλλει έτσι ώστε να επιστρέψουν γρήγορα οι επιβάτες ε, στα σπίτια τους. Γιατί και εκεί είδαμε ότι έχει τα όρια τη αυτή η διαδικασία και αυτή η προσπάθεια. Και τέλος, έχουμε καλή διαχείριση κινδύνου για τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει αυτό το Ινστιτούτο στο Λονδίνο. Μα είναι αυτό για να ενημερώνει για σεισμούς. Και ε, στο περιθώριο και για ηφαίστεια και αυτοί κάνουν προβολές με υπολογιστές. Μα μπορεί αυτό να μας βοηθήσει. Τι, τι κάνουν οι άλλοι, η Αμερική, η Ινδονησία που κάθε τρεις και λίγο εκρήγνεται ε, τα ηφαίστειά τους. Κάνουν άλλες ε, μετρήσεις, είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, κάτι τέτοιο ακούω. Στην Ευρώπη δεν το περιμέναμε. Ωραία, δεν το περιμέναμε, αλλά τώρα κάτι να κάνουμε. Είμαστε πολύ ε, ε προηγμένοι τεχνολογικά, έχουμε μεγάλες δυνατότητες και οι ερευνητές στη Γερμανία έχουν ζητήσει ένα ειδικό δίκτυο ε, ε, μέτρησης ε, της τέφρας, της ποδού και να δούμε λοιπόν πώς θα βελτιώσουμε την τεχνική μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μέσνερ. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ τώρα για δύο λεπτά εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ έκλεισε ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος και αυτό ήταν αναμφίβολα ένα προληπτικό μέτρο ασφαλείας απαραίτητο. Εκ των υστέρων τώρα και πριν ε, κλείσει για δεύτερη φορά εναέριος χώρος, κανονικά θα πρέπει να έχουμε μια πιο καλή ε, αντιμετώπιση του προβλήματος. Και φοβούμε ότι δυστυχώς έχουμε αποτύχει ικτρά και στο συντονισμό και στις μετρήσεις και στην αξιολόγησή τους και ε, στο πώς αντιμετωπίζουμε τους επιβάτες. Και τη δεύτερη φορά η μεταχείριση των επιβατών που περιμέναν τις πτήσεις τους που ε, έπρεπε να διοχετευτούν αλλού, ε, η πληροφόρηση τους ήταν πάρα πολύ ελληματική. Πρέπει να βελτιωθεί οπωσδήποτε αυτό. Διερωτώ με πότε θα έχουμε σχέδια έγκυρα. Κύριε Πίτροπε, ε, μιλήσατε για τα οικονομικά και για τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά δεν τα απαντήσατε με μεγάλη σαφήνεια για να το πω έτσι. Αλλά ε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό, επίκαιρο και απασχολεί συνέχεια τον κόσμο. Πώς θα λυθεί αυτό άραγε, ποιος θα πρέπει να αποζημιωθεί, οι αεροπορικές εταιρείες, θα δώσουν τα χρήματα στους επιβάτες. Επιχειρηματίες που έχασαν σημαντικά ραντεβού θα αποζημιωθούν. Η εταιρεία που περιμένει τα ανταλλακτικά θα αποζημιωθεί. Γιατί μόνο οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν το θεωρώ δικαιολογημένο αυτό, αν το συγκρίνουμε με τις οικονομικές επιπτώσεις που είχε η ιστορία αυτή και η κρίση σε όλο τον κόσμο. Επίσης, έχουν μόνιμη επιδότηση οι αεροπορικές εταιρείες αφού δεν πληρώνουν φόρο για την κυροζήνη. Έχουν πάγια επιδότηση από την αρχή με τη φορολογική αυτή ελάφρυνση. Λοιπόν, επίκειται αυτό το ερώτημα κύριε Επίτροπε και περιμένω να μου απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Λιχτεμπέρκερ. Ο κύριος Ζήλε έχει το λόγο τώρα από τους Ευρωπαίους συντηρητικού και Μεταρρυθμιστές. Κύριε ε, ε, Πρόεδρε, Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κάλλας για όλα όσα έκανε τις τελευταίες πέντε ημέρες. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο-τρεις πρώτες ημέρες ήταν και ό,τι καλύτερο από πλευράς ε, δράσης, αλλά νομίζω ότι μετά έκανε πολύ καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, οι αποφάσεις του Συμβουλίου και σε σχέση με τα λειτουργικά τμήματα ένα αέριου χώρου και σε σχέση με την πρωτοβουλία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και τα περισσότερα μέτρα. Νομίζω ότι όλα αυτά έγιναν εγκαίρως. Θα πρέπει βέβαια ταυτόχρονα να καταλάβουμε τις πολύ μεγάλες πιέσεις που ασκήθηκαν από τους πολιτικούς, από τους και τα δικαιώματά τους, αλλά και από τι αεροπορικές εταιρείες. Πρέπει να δούμε λοιπόν και την νομική βάση, πρέπει να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του ανοίγματο του κλεισίματος του εναέριου χώρου. Φανταστείτε να είχε γίνει ένα ατύχημα λόγω της εφαστιακή τέφρα. Αν η Κομισιόν είχε λάβει τη λάθο απόφαση, για σκεφτείτε τι θα γινόταν. Τότε δεν θα μιλούσαμε για κάποιες απώλειες. Θα μιλούσαμε πλέον για ευθύνες, για καταλογισμό ευθυνών θα ήταν τελώς διαφορετικά τα πράγματα. Επομένως, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και αυτό θα πρέπει να γίνει ε, με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Λήφθησαν κάποιε βραχυπρόθεσμε αποφάσει. Ο κ. Αλχαντραού είπε και για τα δικαιώματα των επιβατών, είπε και για τι αεροπορικέ εταιρείε. Ε, κάποιε εταιρείε δεν ε, σεβάστηκαν τα δικαιώματα των επιβατών τους. Δεν μιλάμε για τρίτες εταιρείε, μιλάμε για αεροπορικέ εταιρείε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκατέλειψαν τους επιβάλλοντες τους και ουσιαστικά ασχολούνταν μόνο με τα χρήματά τους. Πρέπει να δούμε το θέμα λοιπόν, είναι πρόκληση αυτό, το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών. Μια άλλη πρόκληση είναι και το ότι δεν υπάρχει ε, σωστή διασύνδεση των μεταφορών. Ευχαριστώ. θα μιλήσει τώρα για 1,5 ε, λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και άλλες, πρέπει να επικρατήσει η αρχή της προφύλαξης, όπως και οποτεδήποτε διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε ακραίες αποφάσεις που... Ε, θα πρέπει να, που θα στρέψουν τους πολίτες κατά της αρχής της προφύλαξης. Ένα αρχαίο μοντέλο μετεωρολογικό επικράτησε και όχι η γνώμη των πιλότων που ήθελαν ε, να κάνουν ε, δοκιμαστικές πτήσεις. Και ακολούθησε όλη αυτή η αναταραχή στα αεροδρόμια αν διάφοροι ψηλά ιστάμενοι έτυχαν καλής μεταχείρισης, μεγάλος αριθμός πολιτών ε, εγκαταλείφθηκε από όλους και από τις κυβερνήσεις τους. Γι' αυτό ζητάω μια ε, επιτροπή έρευνας κοινοβουλευτική που να ε, αποκαλύψει αυτούς τους απαταιώνες που υποφελήθηκαν από μια τέτοια κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα για την Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Συμπράσας για δυόμιση λεπτά παρακαλώ gerbiama Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, οι συνάδελφοι είπαν πολλά πράγματα σχετικά με την ε, ηφαιστειακή έκρηξη και τις συνέπειες που είχε για τους ε, επιβάτες που παγιδεύτηκαν στα αεροδρόμια. Χαίρομαι που οι αποφάσεις ε, σχετικά με την ε, υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ε, προωθούνται και ότι ε, τα λειτουργικά τμήματα ενεργείου χώρου ε, αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις αρχές Μαΐου. Όμως ε, δεν είμαι σίγουρος αν στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε στρατηγικές που θα περιλάμβαναν και εναλλακτικού τρόπους ε, μεταφοράς, όπως ανέφερε ο συνάδελφος από την Γερμανία. Ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, παραδείγματο χάρη, ή να πάρουμε υπόψη μας και τις χώρες της Βαλτικής, στη Βόρεια Ευρώπη. Η φεστιακή τέφρα πραγματικά ε, ανέδειξε την σπουδαιότητα των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών. Ε, καταλαβαίνω ότι παρόμοιε συνθήκε υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, αλλά μιλάω τώρα για την περιοχή της Βαλτικής. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό θα ήταν ε, η, μια λύση. Αν παραδείγματο χάρη, είχαμε μια σιδηροδρομική σύνδεση με την Πολωνία, θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε πρόσβαση στη Δυτική Ευρώπη. Διαφορετικά παραμένουμε ε, αποκομμένοι από το κεντρικό σιδηροδρομικό σύστημα της Ευρώπης ένα σύγχρονο ε, σύστημα ε, σιδηροδρομικών μεταφορών ε, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει στις άλλες χώρες. Στις βαλτικές όμως χώρες δεν έχουμε αναπτυγμένο σύστημα σιδηροδρόμων. Ρωτάω λοιπόν τον Επίτροπο αν υπάρχουν σχέδια να εστιαστεί η προσοχή σε τέτοιου είδους εναλλακτικά σχέδια μεταφορών. Ξέρω ότι θα χρειαστεί, η, ε, θα χρειαστεί μεγάλη πολιτική βούληση για να αποφύγουμε παρόμοια προβλήματα σε μελλοντικέ κρίσεις. Πασκουάλ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Κάλλας, για τη δουλειά σας αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η συζήτηση αυτή είναι αναπόφευκτη, αγαπητοί συνάδελφοι, και δυστυχώς ε, είναι και αόριστη. Δηλαδή, θα τα ξαναδούμε αυτά τα μαύρα στοιχεία της ε, κατάστασης αυτής και ε, τις στην οικονομία. Αρκεί να θυμίσουμε ποιοι επλήγησαν. Οι ε, επιβάτες, 10 εκατομμύρια, χωρίς ε, οδηγίες τι να κάνουν και χωρίς πτήση. Εντάξει οι οδηγίες και οι κανονισμοί, ποια είναι τα δικαιώματα των ε, ε επιβατών. Σου λέει άλλο είναι θεομηνία, είναι ανωτέρα βία. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο που να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες, η ΆΤΑ υπολογίζει ότι χάσανε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 850 εκατομμύρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο λέει η Ευρωπαϊκή ε, ε υπηρεσία. Η κρίση καλπάζει και απειλούνται πολλές εταιρείε να κλείσουν. Άλλο που επλήγει ο τουρισμός. Ήταν καταστροφικέ οι συνέπειε γιατί ε, ακυρώθηκαν και συμβάσει, ε, αυτές που γίνονται εκ των προτέρων ε, συνήθως για το καλοκαίρι. Και επίση η ανασφάλεια ε, οδήγησε και σε αλλαγή ε, του τρόπου με τον οποίο συνάπτονται οι συμβάσει για την τουριστική περίοδο. Το συμπέρασμα μονοσήμαντο. Δεν έχουμε ε, κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τέτοια κρίση με τρόπο σωστό και κριτική. Γιατί η κριτική είναι απαραίτητη και αναπόφευτη. και αυτοκριτική αν θέλετε. Ε, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις χείρες μας. Όλοι οι φορείς άργησαν να δράσουν, έδρασαν αναποτελεσματικά ε, και με κακό τρόπο. Τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα, τέσσερις ολόκληρες μέρες έκαναν να αντιδράσουν και έβαλαν ως ύψιστο αγαθό την ασφάλεια. Αλλά αυτό ε, δεν οδήγησε σε καθησυχασμό του ε, κόσμου, αλλά σε παράλυση. Τι μέτρα χρειάζονται. Είναι καλά τα μέτρα αυτά που λέτε, αλλά θα πρέπει να είναι και πιο συγκεκριμένα στην εξέλιξή τους. Και δεν το έχουμε ξεχάσει. Σήμερα παραμένει ε, η απειλή. και αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι εξαρτώμαστε από τα ρεύματα του ανέμου και τι διεύθυνση θα πάρει. Και αυτό το είχε πει κάποιος μεγάλος ε, ε, Ισπανός ναυτικός για μια ναυμαχία που χάσαμε. Ε, δεν θα πρέπει εμείς να δείχνουμε τσιγκουνιά τώρα στα μέτρα που θα πάρουμε. Θα μας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά το ηφαίστειο. Ε, ζητώ συντονισμό και ταχεία λήψη αποφάσεων. Να είμαστε ε, γενναιόδοροι ε, και να σκεφτόμαστε εναλλακτικέ λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ε, εγώ δεν λέω ότι φταίει ούτε το Συμβούλιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να κάνουμε τη διάγνωση ότι δεν καταφέραμε να λύσουμε και αυτή την κρίση τέτοια διάσταση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κάλεσα για την δράση του όλε αυτέ τι ημέρε και να πω ότι αυτή η κρίση στην κινητικότητα λόγω τη βαστιακή τέφα που και χθε είχε ω αποτέλεσμα να κλείσουν ε, ε, εναέροι χώροι τη Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε και κάποιε συνεδριάσει βέβαια που συγκάλεσε η Ισπανική Προεδρία. Πολλά πράγματα μας έχουν διδάξει. Πρώτα απ' όλα ότι επλήγει όλο ο κλάδο, όχι μόνο αεροπορικές εταιρείε, τα ε, αεροδρόμια και γι' αυτό επικροτούμε που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ό,τι αφορά τι βοήθειε και τι αποζημιώσει. Ε, ο κύριο Κάλλο, ο κύριο ε, Σαλμούνι και ο κύριο Ταγιάννη. Ε, θα χαιρετήσουμε λοιπόν την πολύ σωστή προσέγγιση και εστίαση του θέματο από την Κομισιόν. Είναι απαραίτητο ο νέο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Πλέον ξέρουμε ότι είναι και κατεπήγον να, να ισχύσει αυτή η πρωτοβουλία και θα πρέπει να έρθουν τα εμπόδια που υπάρχουν έχουν στο Συμβούλιο. Θα πρέπει επίση να δρομολογηθεί και να είναι εγγυημένη και η χρηματοδότηση του προγράμματο ΣΕΖΑΡ. Θα μπορούσε να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχουν και ποιε είναι αυτέ οι δυσπιστίε, οι καχυποψίε που εκφράστηκαν στο Συμβούλιο τη 4η Μαου. Θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Και ποια είναι τα ε, κράτη τα οποία άλλοι ανοίγουν λιγότερο, άλλα περισσότερο. Αυτό δεν είναι καλό για τον ανταγωνιστικό, τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπαμε για τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Βλέπουμε ότι θα πρέπει να, δούμε, ε, να αναθεωρήσουμε την εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρή, άτεγκτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, βλέπουμε ότι κάποιε εταιρείε είπαν ψέματα στου επιβάτε και δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να τιμωρηθούν. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Εμεί ω πολιτική ομάδα το είχαμε προτείνει για τον προπολογισμό του 2010 να υπάρχουν ε, ε, ε, γραφεία ενώσεων καταναλωτών στα αεροδρόμια για να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και να υιοθετούνται τα κατάλληλα μέτρα για τους καταναλωτές και για τους επιβάτες. Εμείς βέβαια είμαστε και υπέρ των ευρωπαϊκών δικτύων, των συνδεσμένων μεταφορών, με το σιδηρόδρομο. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες επιπτώσεων, είδαμε με τη διασύνδεση Βαρκελόνης Μαδρίτης. Πρέπει πραγματικά να υπάρξει ένα εναλλακτικό δευτερεύον σύστημα κινητικό όπως αυτό που γίνεται στον τομέα του ηλεκτρισμού και των τηλεπικοινωνιών και θα πρέπει να δούμε και τις δημοσιονομικές προοπτικές να είναι πιο φιλόδοξες στο τομέα των ε, ευρωπαϊκών. Το χρόνο, και κύριοι συνάδελφοι. Η κυρία Χόρκιν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Thank you, Madam President. My particular perspective... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ενδιαφέρομαι περισσότερο για τα πιο περιφερειακά αεροδρόμια, και τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν ήδη ε, οικονομικές δυσκολίες. Ζω σε ένα νησί και οι τύχοι των περιφερειακών αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών έχουν μεγάλη σημασία. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, διάφορα αεροδρόμια στη δική ακτή της Ιρλανδίας. Και πρέπει να καταλάβετε ότι λόγω τη ε, γειτονική μας θέση με την Ισλανδία έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με την ΤΕΦΡΑ. Για τα περιφερειακά αεροδρόμια ε, πιστεύω ότι η ε, Κομισιόν θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα μέτρα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν πραγματική ευελιξία ε, όσον αφορά την κατάσταση των περιφερειακών αεροδρομίων. Από την άλλη μεριά υπάρχουν αεροπορικέ εταιρείε που έχουν ήδη οικονομικά προβλήματα και μπορεί να χρειαστεί να σταματήσουν τι δραστηριότητέ του λόγω αυτή τη κρίση. Αν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα, αυτό θα οδηγήσει σε απώλειε θέσει εργασία και σε λιγότερο ανταγωνισμό στην αγορά. Πρέπει λοιπόν η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο και μέσω μιας δίκαιης κατανομής της οικονομικής βοήθειας και ε, με άλλα μέτρα που διαθέτει. Τέλος, θα πρέπει να ε, ληφθούν νομοθετικά μέτρα ε, ώστε να μην μπορούν οι αεροπορικές εταιρείες να καταργούν τις πτήσεις τους διότι ε, οι συνέπειε είναι σημαντικέ για όλου, για του επιβάτε, για τα αεροδρόμια, για τι αεροπορικέ εταιρείε. Το θέμα είναι ποιο είναι υπεύθυνο και ποιο ε, φέρει το οικονομικό βάρο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, προτείνεται ένα σύστημα διαχείριση και συντονισμού τη κρίση, Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη και ξαναζούμε τα ίδια προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να πω, όπως και άλλοι, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι διαλειτουργικά τα συστήματα κρατήσεων για το σιδηρόδρομο. Θα πρέπει οι χερσαίες μεταφορές και ο σιδηρόδρομος να γίνεται πιο εύκολα και να αντικαθιστά ε, τα αεροπλάνα όταν έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα ηφαίστεια, μπορεί να υπάρξουν και άλλες καταστάσεις που να μπλοκάρουν τις αερομεταφορές. Ε, κάτι άλλο όμως πιο διαρθρωτικό, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για την κάλυψη του κινδύνου ε, από τον ίδιο το κλάδο, από τον ίδιο το κλάδο επιμένω σε τέτοιου είδου περιπτώσει. Γιατί πιστεύω ότι οι κρατικές ενισχύσεις κάθε φορά που δίδονται ή που υπάρχει πρόβλημα, πολύ γρήγορα θα είναι αφόρητε από πλευρά δημοσιονομική Και είναι και τεράστιες οι διακρίσει μεταξύ των εταιριών ε, ε, από χώρα σε χώρα. Και κάποιοι θα ήταν δικαιούχοι και κάποιοι θα αποκλείονται. Ακριβώ επειδή έχουν μεγάλο βάρο οι εταιρείε, θα πρέπει να έχουμε ε, όπως και στις τράπεζες, ε, ένα σύστημα φρόνησης ε, και συνετής ε, διαχείρισης με ένα σύστημα ασφαλίσεων και ατασφαλίσεων όπως υπάρχουν στις τράπεζες για να μην ζητάμε από τα κράτη δωρεάν να ασφαλίζουν τις εταιρείες που έτσι και αλλιώς για ιστορικούς λόγους δεν πληρώνουν φόρο στις κυροζήνη. Και θα πρέπει οι εταιρείε να αποζημιώνουν όπως πρέπει τους ε, καταναλωτέ, χωρίς να πληρώνουν γι' αυτό οι φορολογούμενοι όμω. Για τρία λεπτά. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, όλοι καταλαβαίνουμε τις τεράστιες διαταραχές που προκλήθηκαν και συνεχίζουν να προκαλούνται από το σύννεφό της ηφαιστιακής τέφρας. Πάνω από 100.000 ε, ακυρώθηκαν και 12 εκατομμύρια επιβάτε δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν σύμφωνα με τα σχέδιά τους. Εμπορεύματα ε, καθυστέρησαν ή δεν μεταφέρθηκαν καθόλου και οι επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες επηρεάστηκαν και όλες οι αεροπορικές εταιρείε και τα αεροδρόμια της ε, Ευρώπη υπέστησαν καταστροφικέ οικονομικέ απώλειες. Ε, σε όλο αυτό το χάος ένα πράγμα είναι σαφές, ότι οι αεροπορικές μεταφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομία και ως άτομα εξα, εξαρτόμαστε από μια ευημερούσα ε, ε, βιομηχανία αεροπορικών μεταφορών, όπως και η ασφάλιση σε εξαρτάται από αυτό. Ε, χαιρετίζουμε την αποφασιστική απάντηση που έδωσε η Κομισιόν ε, η Κομισιόν αναγνώρισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι οικονομικές αποζημιώσεις αλλά επίσης και η ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων ΣΕΖΑΡ. Γενικά, ο κανόνα πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ότι το κράτο δεν θα πρέπει να υποστηρίζει τι επιχειρήσει, διότι το ρίσκο είναι μέρο τη επιχειρηματικότητα. Όμω, σε εξαιρετικέ συνθήκε, ε, όταν υπάρχουν τόσο τεράστιες οικονομικές απώλειες, ε, όπως κατά την 11η ε, Σεπτεμβρίου, ε, θα έλεγα τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν μέτρα ενίσχυσης του, του κλάδου. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για να αντιμετωπιστούν τέτοιε κρίσει. Πρώτα απ' όλα, οι αεροπορικέ εταιρείε πρέπει να συμμετέχουν στι συζητήσει σχετικά με ε, το πιθανό κλείσιμο του ενέργειου χώρου εξ αρχή. Δεύτερον, όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται με ένα λογικό τρόπο. Και εξακολουθώ να έχω αμφιβολίε σχετικά με την ε, μέθοδο που ακολουθήθηκε. Ε, Παραδείγματο χάρη, ποιο θα ήταν ο ακριβή ρόλο του ε, συντονιστή αυτού, του συντονιστικού, ε, του συντονιστή. Ε, υπό ποιε συνθήκε θα εργαζόταν. Θέλω όλα αυτά να τα εξετάσουμε λεπτομερώς κύριε Επίτροπε πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία. Διότι μια βιαστική απάντηση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά. Επίσης να δούμε τι κάνουν στη Βόρεια Αμερική και αλλού στον κόσμο για την αντιμετώπιση της ε, τέφρας. στο Ηνωμένο Βασιλείο χρησιμοποιούν τη μέθοδο αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μια άλλη μέθοδο για τη μετατόπιση της τέφρας. Πρέπει να ε, δούμε τι κάνουν και εκεί. Επίσης, οι συνέπειες ε, τέτοιων αποφάσεων δεν μένουν εντός των ε, ορίων μας, των συνόρων μας. Πρέπει να δούμε τι κάνουν και οι άλλες χώρες. Και τέλος, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την ευθύνη ε, να αναπτύξουν μια μακρόπνοη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τα θέματα αυτά. Ε, πρέπει να ληφθούν μέτρα για βελτίωση της διαχείρισης, σίγουρα να εφαρμοστούν σχέδια αποζημίωσης χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και καλά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το κλείσιμο του ενέργου χώρου μετά την ε, έκρηξη του Ισλανδικού ηφαιστείου τον Απρίλιο επιβεβαίωσε την, ε, το πόσο ευάλωτε είναι στι ε, φυσικέ συνθήκε οι ενέργειε μεταφορέ. Και δεν μιλάμε μόνο τώρα για την έκρηξη ηφαιστείου, μιλάμε για την ομίχλη, για τι ισχυρέ βροχοπτώσει, χιονοπτώσει, ανέμου που δημιουργούν προβλήματα στι τακτικέ πτήσει των αεροπορικών εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν οι υπεύθυνε αεροπορικές εταιρείες ε, συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, συνάπτουν ασφαλίσεις για να καλυφθούν ε, προβλήματα που προκύπτουν από τέτοιους αστάθμιτους παράγοντες. Και βέβαια το κόστος της ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται στο εισιτήριο το εμπορικό που πληρώνουν οι επιβάτες. Και πολλές φορές και στα εισιτήρια ε, προβλέπεται και η παροχή βοήθειας για περίπτωση κάποιου έκτακτου συμβάντος. Θέλω να επαναλάβω το εξή, κύριε Επιτροπή. Ορισμένοι επιβάτε πληρώνουν όταν αγοράζουν το εισιτήριο, πληρώνουν την εταιρεία για να λάβουν επαναλαμβάνω, βοήθεια σε περίπτωση κάποιου έκτακτου γεγονότος και μετά ε, τους αποζημιώνουν οι ασφαλιστές τους, τους τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν χρησιμοποιεί Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο και να αποζημιώσει όλους αυτούς που έχουν υποβάλει αυτά τα αιτήματα και δεν θέλει τελικά γι' αυτό το λόγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ικανοποιήσει όλα αυτά τα αιτήματα. Αν ε, επιβληθούν λοιπόν κάποια, κάποιοι περιορισμοί θα πρέπει οι ασφαλιστικοί φορείς να καταβάλουν τις αποζημιώσεις έτσι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν υπάρξει φωτιά ε, στο σπίτι, αν υπάρξει, ε, πέσει στέγη και αν είναι ασφαλισμένο το σπίτι, καλύπτεται ο ασφαλισμένος. Ε. Δεν θα μπει η κυβέρνηση για να προσφέρει ένα καινούριο σπίτι ή να επισκευάσει το σπίτι. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τι απώλειε των αεροπορικών εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πεπισμένο ότι σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον δεν υπάρχει καμία δυνατή αιτιολογία για υποστήριξη ουδήποτε είδους προς αεροπορικές εταιρείες από τις κυβερνήσεις και επομένως τελικά από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το λόγο θα πάρει για τρία λεπτά η κυρία Σκριντλεύσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, τον Απρίλιο ξεράγει το ηφαίστειο και παρέλυσε πλήρως ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι ανωτέρα βία, αλλά είχε τρομερές ε, συνέπειες για τους επιβάτες και τις αεροπορικές εταιρείες. Σε δεκάδες αεροδρόμια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένοι, αποκλεισμένοι επιβάτες χωρίς να έχουν καμία πληροφόρηση. Με ε, μοναδικές εξαιρέσεις ε, ε, και οι μόνες αξιόπιστες προφορίες ήταν ποια αεροδρόμια κλείνουν ακόμα και τίποτα άλλο. Βεβαίως ε, δεν φταίει κανείς για αυτή την κατάσταση, είναι φυσική καταστροφή, η θεομηνία, αλλά ε, πώς συμπεριφέρθηκαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θεσμοί που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια των επιβατών. Τα μέτρα ήταν και ανεπαρκή και καθυστερημένα. Ε, χάος τεράστιο επικράτησε και τεράστια ανασφάλεια για το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, αυτό ε, είναι αρνητικό ως γεγονός και θα ήθελα να ρωτήσω τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον, σε περίπτωση που συνεχίζει να εκρήγνεται το υφέστη αυτό. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται σωστά μια τέτοια κατάσταση και με πρόληψη και τι προτίθεται να κάνει για την ενημέρωση και το καθήκον που έχει να ενημερώνει τους ε, επιβάτες. Νομίζω ότι τα μέτρα που έχετε προτείνει έως τώρα είναι επαρκή. Κύριο Δανέλη, θα πάρει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το κλείσιμο δύο σημαντικών ευρωπαϊκών αερολιμένων χθε στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ λόγω νέα ισόρευσης ηφαιστειακής τέφρας κατέδειξε ότι η καθήλωση πτήσεων τον Απρίλιο δεν ήταν αποτέλεσμα ενός απίθανου συμβάντος άνευ μακροχρόνιων επιπτώσεων ή κινδύνου επανάληψης. η απουσία εξάλλου του συναδέλφου Σίμψον απόψε από τη συζήτησή μας είναι πολύ πιο ηχηρή από την παρουσία του. διανύουμε μια δύσκολη οικονομική περίοδο που φέρνει απανοτές συγχωνεύσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και που διέπεται από αβεβαιότητες ε, για τις εταιρείες αλλά και τους εργαζομένους αυτών. Για τρεις συνεχόμενες μέρες τον Απρίλιο οι καθημερινές απώλειες του διεθνούς κλάδου έφτασαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των οικονομικά ασθενέστερων αερομεταφορέων της Ευρώπης. Είναι βέβαιο ότι έλειψαν και συνεχίζουν να λείπουν τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία που να επιτρέπουν η αξιολόγηση ρίσκου να λαμβάνει η χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αξιοποιεί βάσει συγκεκριμένης μεθόδου όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκές αρχές. ο κίνδυνος επανάληψης της εξαιρετικά επιζήμιας σύγχυσης που ζήσαμε κάτω από τις στάθειε του ηφαιστείου είναι υπαρκτός και πρέπει τα μέτρα που θα πάρθουν να θωρακίζουν θεσμικά την ικανότητα της ένωσης να παρεμβαίνει με συντονισμένο και προμελετημένο τρόπο σε κρίσει αυτού του είδους περιορίζοντας την απίστευτη ταλαιπωρία εκατομμυρίων επιβατών και την οικονομική ζημιά αερομεταφορέων και τουριστικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δανέλη. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Γκάλαγκερ για 1,5 λεπτό. Uh, does not have a land uh, connection to mainland Europe. Η Ιρλανδία δεν συνδέεται χερσαία με την Ευρώπη και οι Ιρλανδοί επιβάτες γνώρισαν τεράστια προβλήματα και τολμώ να πω περισσότερο από άλλα κράτη-μέλη. Εγώ ο ίδιος παράδειγμα που ήρθα στο Στρασβούργο ε, χρειάστηκε να πάρω ferry boat για την Ουαλία και μετά ε, άλλο ferry boat για τη Γαλλία και τρένο για το Στρασβούργο. Το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό για αυτό που κάνουν και αυτά που τραβάνε οι Ιρλανδοί ε, τις τελευταίες εβδομάδες. Οι Υπουργοί Μεταφορών ε, κάνουν ε, προσπάθειες για ειδικά μέτρα, αλλά πρέπει να πω ότι πάνω από 300.000 ε, ώρες πτήσεων έχουν γίνει. Βεβαίως είναι καλό αυτό και χρειάζονται και άλλα μέτρα. Ε, υποστηρίζω τα μέτρα για ταχεία υιοθέτηση ε, της έννοιας του ενιαίου ευρωπαϊκού ε, ουρανού. Το Φεβρουάριο στη Μαδρίτη η Ισπανική Προεδρία έλαβε μια απόφαση που ε, δρομολογεί αυτή την εξέλιξη και ελπίζω, χαίρομαι που είναι εδώ ο Επίτροπος. Είναι χμή του δόρατο στην προσπάθεια αυτή. Και επίση να δούμε και το ρόλο του Eurocontrol και να το εξετάσουμε πολύ στενά. Θα πρέπει ε, να έχει και δυνατότητες ουσιαστικές, όχι μόνο συντονιστικές όπως έχει αυτό τον καιρό. Ε, τώρα είδαμε ότι η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είδαν την ενέργεια κυκλοφορία τους να διαταράσσεται. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να έχει σύνορα ούτε πολιτικά ούτε γεωγραφικά αλλά ήρθε το ηφαίστειο να μας θυμίσει ότι η φύση βάζει όρια. Και χρειάζεται μια κοινή πολιτική στην Ευρώπη ε, και ένα ενιαίος ουρανό. Βολτσίτης έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Κρατήστε το χρόνο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι συνέπειε τη ηφαιστιακή έκρηξη έχουν γίνει αισθητέ στα συστήματα αερομεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη ακυρώθηκαν πάνω από 100.000 πτήσεις και τι συνέπειες τις ένιωσαν πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Οι συνέπειες αυτές ε, ήταν ιδιαίτερα πιο ε, σοβαρές για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, που είναι απομονωμένες, αποκομμένες, δεν έχουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε καλύτερα διευρωπαϊκά ε, μεταφορικά δίκτυα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό για τη μεταφορά και των εμπορευμάτων και των επιβατών. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό ε, σύστημα λοιπόν που να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις ε, αερομεταφορές. Πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα άλλα μέσα μεταφοράς, ιδίως για μέσα στην Ευρώπη. Ε, πρέπει να υπάρξει ένα καλό σύστημα με καλές διασυνδέσεις που θα ωφελήσει και τους επιβάτες και την λειτουργία της οικονομίας μας. Επίσης υποστηρίζω την ιδέα να υπάρξουν πρόσθετες διασυνδέσεις ε, αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους σιδηροδρομικούς διαδρόμους και δημιουργία τέτοιων διαδρόμων στην Ευρώπη και επιπλέον ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάτι τέτοιο θα έχει πρόσθετη αξία για ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, θα πάρουν το λόγο συνάδελφοι για ένα λεπτό. Προσέξτε να μην το ξεπεράσετε σας παρακαλώ. Πρώτος ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για τον τουρισμό. Ένα πολύ σημαντικό τομέα για τα Κανάρια νησιά που υποδέχονται 12 εκατομμύρια τουρίστες στον κόσμο. Αυτό το οποίο χρειάζονται οι τουρίστες είναι βεβαιότητα αυτά τα φαινόμενα και αν υπάρχει περίπτωση να επαναληφθούν ε, έχουν δραματικές επιπτώσεις για το στρατηγικό τομέα για τα Κανάρια νησιά. Και είχαμε επιπτώσεις όχι μόνο για τα, ε, για τα αεροδρόμια και για τις οροπορικέ εταιρείε, αλλά για τον τομέα της εστίας, των ξενοδοχείων, των μεταφορών, ε, όλοι. Από τις 15 έως τις 30... Ε, Απριλίου Είχαμε 57,3 εκατομμύρια ευρώ απώλειες ε, γενικότερα στην περιοχή μου και καταλαβαίνετε ότι το νυχτερινό άνοιγμα ε, των ε, ανανοιχτά, δηλαδή τη νύχτα τα αεροδρόμια για να παραμείνουν εκεί οι επιβάτες αλλά και οι απαραίτητες υπηρεσίες προς τους επιβάτες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια πρέπει να προσέξουμε να αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Αγαπητέ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το στένο σας, για την ασφάλεια των επιβατών. Τις τελευταίες ημέρες είδαμε ότι η κερδοσκοπία δεν είναι μόνο στο χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και στην ασφάλεια των επιβατών ορισμένη. Και είναι πολύ γενναιόδορη, ευτυχώς μόνο στα λόγια προς το παρόν και όχι στα έργα. Και το θέμα δεν είναι μόνο οι επιβάτες ε, των ε, αεροπλάνων που κυκλοφορούν στον αέρα, αλλά και οι άλλοι που ζουν στη γη. Και σας ενθαρρύνω να προχωρήσετε στην ίδια κατεύθυνση. Τι γίνεται με τα δικαιώματα των επιβατών. Μάθαμε πρόσφατα ότι δεν έχουν όλοι ε, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε όλες οι ηλικίε. Και είχαν μπλοκαριστεί τα τηλέφωνα, δεν υπήρχε επικοινωνία ε, και δεν είναι και ο κόσμος συνηθισμένος κάθε μέρα να κυκλοφορεί όπως εμείς ε, οι επιχειρηματίες ε, με αεροπλάνα. Οι τουρίστες που πετάνε σπάνια, οι ηλικιωμένοι είχαν πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ σας να να ακολουθήσετε την έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση η οποία προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Ισλανδίας δείχνει πόσο σημαντικό είναι ο αντίκτυπος ορισμένων φυσικών φαινομένων που ευτυχώ είναι σπάνια. Αλλά αν ε, επαναληφθούν ε, δημιουργούν ε, προβλήματα και διαταραχές και γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια προληπτική προσέγγιση στην περίπτωση αυτή βέβαια όχι να προλάβουμε γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν αλλά να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε να προσαρμόσουμε σε έφτατο χρόνο και να υιοθετήσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειωθεί ο αντίκτυπο αυτών των καταστροφών. Ωστόσο δεν θα πρέπει να γίνονται, να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες με υποτιθέμενο στόχο την ασφάλεια, ενώ άλλοι είναι οι στόχοι επιδιωκόμενοι. Παραδείγματο χάρη η απελευθέρωση τη ε, ε, εναέρεια κυκλοφορίας και των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη. Αν κάτι επιβεβαιώθηκε στην, με την κρίση αυτή είναι ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτερε προσπάθειες στη διαχείριση τη αεροπορική μεταφορά και να, θα πρέπει να δούμε υπέρ, ε, υπέρ των πολιτών και να μειώσουμε την ασφάλεια. Το παρακαλώ. Κύριε ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπη, μιλούμε για τις διαταραχές στην ενέργεια κυκλοφορία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Θέλω όμως να το λύσω εγώ την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι το ύψιστο αγαθό. Κύριε Επίτροπε, κάνατε πολλά βήματα. Έχει έρθει η ώρα τώρα συγκεκριμένα να προτείνουμε εναλλακτικέ λύσεις και να τις εφαρμόσουμε. Για παράδειγμα, διευρωπαϊκό δίκτυο τρένου υψηλής ταχύτητας και αυτό συμβάλλει στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Σας ευχαριστώ. Το πολύ κύριε Βέρτμαν. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό. Παγκόσμια Έχουμε 2.000 ηφαίστεια και σε έκρηξη και σε ενεργή φάση αυτή τη στιγμή 50. Δεν είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, είναι διεθνές. Και εδώ θα πρέπει η έρευνα να μας βοηθήσει και να μας εξηγήσει πού είναι η πραγματική κίνδυνη και πού ε, υπάρχει η ευθύνη και πόσο ευρεία είναι αυτή. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον Επίτροπο να το κοιτάξει μαζί με το Eurocontrol και να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα να κάνει έρευνα ακριβώ για να αξιολογεί σωστά το κίνδυνο. Γιατί ε, σε τελική ανάλυση ο κυβερνήτη ενό αεροσκάφου φέρει την ευθύνη, ε, αλλά ε, καλείται και ο καταναλωτή να σκεφτεί αν είναι ρίσκο ή όχι και δεν είναι καθένα υποχρεωμένο να πετάξει. Μπορεί να επιλέξει να πει ότι εγώ δεν παίρνω το αεροπλάνο αν θεωρεί ότι είναι κίνδυνο. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριο ο, κύριος Σκέλη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Σόνο Κέισι είπε ότι όλος ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση χάος. Αν κοιτάξουμε κάτω, βλέπουμε ρήπανση του περιβάλλοντος, αν δούμε προς τα πάνω, βλέπουμε την τέφρα του ε, ηφαιστείου και αν κοιτάξουμε αλλού, βλέπουμε την ύφεση που αποδεκατίζει την οικονομία. Σίγουρα η Ιρλανδία ε, πλήχθηκε περισσότερο από την ε, ηφαιστειακή τέφρα και εγώ δεν μπόρεσα να πάω στις ε, Βρυξέλλες, την άλλη φορά δεν μπόρεσα να έρθω εδώ. Πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι είναι αδύνατο να βρει κανείς ειδηρίο στο Eurostar. Χρειάζεται κανείς πιστοτική κάρτα για να κάνει την κράτηση ε, και αυτό ε, είναι αδύνατον να το κάνει κανείς όταν είναι transit. πρέπει να κάνουμε το ίδιο, ένα ίδιο σύστημα για τα ferry boat για τις αεροπορικές εταιρείες. Διότι έχει μιλήσει ήδη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι μοναδική, αλλά ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να προσθέσω μόνο ότι χρειάζεται κάθε τεχνολογία που έχουμε για να μετράμε ε, την τέφρα. Εγώ πήγα στην Άσπρια στην Τουλούζη ε, και μας ε, είπαν ότι υπάρχει ένα λεπτομερέστατο σύστημα για να μετράνε τα σωματίδια αυτά και με δορυφόρους και δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκε αυτό ε, είναι η ΕΑΝΤΑΕΣ, Ευρωπαϊκή Εταιρεία που τα κάνει αυτά. Κύριε Πίτροπε, το έχετε χρησιμοποιήσει, σκέφτεστε να το χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα. Ολοκληρώσαμε εδώ τις παρεμβάσεις των βουλευτών και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Επίτροπος για να κλείσει τη συζήτηση. members. Αξι... Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, ε, κυρία ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο ενδιαφέροντα ε, σχόλια που κάνετε για το θέμα της φεστιακής τέφρας. Βεβαίως, στην αρχή είχα μόνο τρία λεπτά στη διάθεσή μου και άρα τώρα μπορώ να δεκαπλασιάσω τον χρόνο αν χρειαστεί, αν μπορούσα για όλα αυτά τα θέματα. Θα είμαι σύντομος όμως, δεν θα μακρηγορήσω. Πρέπει μόνο να πω ότι ξέρετε ότι πραγματικά αυτή η περίοδος ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ε, ε, οι συνθήκες πραγματικά ήταν έκτακτες. Είναι γεγονός ότι τα ηφαίστεια μπορούν να ξαναεκραγούν και το Ισλανδικό ηφαίστειο ε, ξαναεξεράγει όντως, αλλά αυτό ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ε, τα ηφαίστεια, είναι οι θύελες, οι χιονοθύελες, όλων των ειδών τα πράγματα που συμβαίνουν και που όλα αυτά μπορούν να αναστατώσουν ε, τις ε, μεταφορές. Αυτό είναι ε, ένας κίνδυνος που κανείς δεν μπορεί να τον λάβει από μόνος του. Ούτε αεροπορικές εταιρείες, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα για την ρύθμιση των αερομεταφορών. Όλα αυτά ε, τα ρυθμίζουν ε, διακυβερνητικοί ε, φορείς και εθνικές αρχές. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πω ότι το να αποκλείσει κανείς, να προλάβει ή να εμποδίσει όλα αυτά που μπορούν να συμβούν στις αερομεταφορές είναι αδύνατον. Και τον κίνδυνο πρέπει να τον μοιραστούμε. Και οι πελάτες που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των αερομεταφορών. Όλοι ε, είμαστε διατεθειμένοι να ε, δεχτούμε κάποια καθυστέρηση γιατί το αεροδρόμιο των Βρυξελών ας πούμε έχει κλείσει λόγω ε, χιονόπτωσης. Όλοι δεχόμαστε ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Τώρα, σχετικά με την κριτική του, που λέει ότι η αντίδρασή μας ήταν καθυστερημένη και ανεπαρκής. Μίλησα με το Eurocontrol και ο κίνδυνος της τέφρας είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Και δεν έχουμε ε, την προσδοκία ότι θα βρεθεί μια επιστημονική απάντηση σχετικά με το ποιο είναι το μέγεθος των σωματιδίων που είναι πραγματικά επικίνδυνο ε, για τους κινητήρες. Κανείς δεν θέλει να κάνει αυτή την εκτίμηση και να πει ότι ναι, αυτή η τέφρα πλέον δεν είναι επικίνδυνη για τους κινητήρες. Κανείς δεν θέλει να, αναλάβει αυτή την ευθύνη. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα πράγματα. Και η απόφαση να κλείσουν τα αεροδρόμια ε, ελήφθη ε, αυστηρά σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες και από τα αρμόδια όργανα. Και αν κάποιος ρωτήσει Ποιος είναι τώρα υπεύθυνο για το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Θα σας ε, ρωτούσα με τη σειρά μου ποιος θα ήταν υπεύθυνο αν δεν έκλεινε ο εναέριος χώρος και κάτι συνέβαινε. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν εμείς ή το Eurocontrol ε, Ε, έλαβε τη σχετική απόφαση δεν ήταν εύκολη η απόφαση, ούτε εύκολη η συζήτηση, γιατί η απόφαση αυτή συνεπάγεται ότι αναλαμβάνει κανείς τεράστια ευθύνη για την ασφάλεια και για, τις, ε, για την ασφάλεια ε, των, των αεροπλάνων και των ζώων βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι υπό τι ε, δεδομένε συνθήκες τα πράγματα έγιναν σχετικά γρήγορα. Γιατί φυσικά η έκρηξη του ηφαιστείου ε, είναι κάτι το εντελώς έκτακτο και απρόβλεπτο. Τώρα, για το μέλλον, το βασικό θέμα που αναφέρθηκε από κάποιους είναι τι ε, θα πούμε για την Ιδονησία ή για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί την ευθύνη την έχουν κυρίως οι, πιλότε, οι πιλότοι. Ε, οι πιλότοι μέχρι στιγμής ε, στην Ευρώπη αρνούνται να δεχτούν μια τέτοια ε, καινούρια ευθύνη. Εν τω μεταξύ η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη ε, στη, στον ενέργειο χώρο της Ευρώπης και χρειάζεται και μεγαλύτερη ευελιξία αλλά σε συνδυασμό με σαφέστερα στοιχεία όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους, τις πιθανές απειλές δεν μπορούμε, δεν ξέρω στην Ιδονησία τι κάνουν, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες το σύστημα είναι πολύ απλό. Ο πιλότος αποφασίζει αν θα πετάξει ή όχι. Και το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά πρέπει να πω. Αλλά στην Ευρώπη προφανώς πρέπει ε, πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε μια κοινή προσέγγιση, μια κοινή μεθοδολογία ε, σχετικά με την ε, δυνατότητα αξιολόγησης του κινδύνου. Τώρα, για τους επιβάτες πρέπει να πω ότι εμείς με μεγάλη συνέπεια ε, λέμε ε, σαν Κομισιόν ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Φυσικά η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας είναι και πάλι στα χέρια των κρατών μελών, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ε, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες και τα περισσότερα κρατημέλη το έχουν πάρει αυτό πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Φυσικά υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις, υπάρχουν και κάποια αρνητικά παραδείγματα για τα οποία θα υπάρξουν και συνέπειες, αλλά οι περισσότεροι τα παίρνουν όλα αυτά πολύ στα σοβαρά και θα κάνουμε μια ε, αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας οπότε και θα ε, κάνουμε μια ε, αξιολόγηση του πώς, των ερμηνειών που δόθηκαν στο θέμα αυτό των δικαιωμάτων των επιβατών. Γενικά πάντως πρέπει να πούμε ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των επιβατών και η λογική λέει ότι οι επιβάτες πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες, τη σχετική ε, φροντίδα και βοήθεια και ε, να ε, αναδρομολογείται το ταξίδι τους. Όχι αποζημίωση, δεν είναι αυτή η λέξη που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Φυσικά υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόγραμμα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και για την ε, διαχείριση των αερομεταφορών. Εγώ δεν μπορώ να παραπονεθώ για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, κατά την περίοδο αυτή. Ε, με πολύ συνεργατικό πνεύμα συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και πάρα πολλέ αποφάσεις ελήφθησαν που υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόντουσαν πολύ περισσότερο χρόνο αλλά πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κακή συνεργασία με τα κράτη-μέλη κατά την ε, προπαρασκευή και, την, και, τον, ε, και τη διεξαγωγή αυτού του έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών. Τώρα, για τις οικονομικές συνέπειες. Οι, απλοί, οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί και περιγράφονται σαφέστατα στο έγγραφο το οποίο ε, συνέταξαν ε, οι τρεις ε, επίτροποι, τρεις αρμόδιοι επίτροποι. Και λέει πάρα πολύ σαφώς το έγγραφο αυτό ότι η κρατική ενίσχυση μπορεί να δοθεί αν το κράτος μέλος θεωρήσει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να χορηγηθεί κρατική ενίσχυση σε αεροπορικές εταιρείες που έχουν προβλήματα. Διότι το κόστο των επιβατών βαραίνει την αεροπορική εταιρεία. Αν τώρα η αεροπορική εταιρεία έχει πραγματικά προβλήματα, βρίσκεται σε πραγματικά πολύ άσχημη κατάσταση, τότε μπορεί να δοθεί κρατική ενίσχυση. Αλλά πριν δοθεί η κρατική ε, ενίσχυση πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ προσεκτική ε, εκτίμηση και αξιολόγηση, ώστε να μην προκύψει στρέβλωση της αγοράς και ε, ε, να μην δοθούν αθέμητα πλεονεκτήματα ε, σε κάποιες αεροπορικές εταιρείε. Και αυτός είναι ο φόβος όλων και η προσέγγιση της Κομισιόν και σίγουρα οι υπηρεσίε ανταγωνισμού της Κομισιόν θα εξετάσουν πολύ προσεκτικά ε, κάθε πιθανή ε, χορηγήση κρατική ενίσχυση. Μέχρι στιγμή, από ό,τι ξέρω, κανεί δεν έχει ε, ζητήσει έγκριση για να δοθεί κρατική ενίσχυση. Ε, από ό,τι ξέρουμε οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τέτοια σχέδια για επίγουσες ε, ανάγκες. Όπως είπαν ε, ε, κάποιοι, πρέπει να είναι ασφαλισμένες οι αεροπορικές εταιρείες έναντι τέτοιων έκτακτων συμβάντων ή ειδικά σχέδια. Και Βεβαίως, ε, σαν οικονομολόγος, ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες υπολογισμού των απολειών. Ε, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια δηλαδή στους υπολογισμούς της ζημιάς που προκάλεσε η φεστιακή τέφρα και που μπορεί να υποβληθεί σαν απέτηση αποζημίωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες. Το Συμβούλιο ε, Υπουργών Μεταφορών θα συνεδριάσει εκ νέου για να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα. Ε, τώρα για τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Ε, το θέμα είναι ε, τι μπορούσαν να κάνουν και τι έκαναν πραγματικά οι σιδηρόδρομοι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Ε, ρώτησα και έλαβα πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για πρόσθετα τρένα, ε, υπάρχει το θέμα της διαθεσιμότητας ε, όλων των πληροφοριών ε, βέβαια, των σχετικών πληροφοριών, των ε, δρομολογίων κλπ. Οι πληροφορίες δεν ήταν ικανοποιητικέ που δόθηκαν. Από την άποψη αυτή λοιπόν μπορούν να γίνουν πολλά στο μέλλον. Δηλαδή καλύτερη ενημέρωση να υπάρχει για όλες αυτές τις εναλλακτικέ δυνατότητες. Φυσικά, όταν υπάρχει μια τέτοια κρίση στις αερομεταφορές, ο ε, παραβατρισμός των ε, επιβατών ε, παραμένει στα χέρια των αεροπορικών εταιριών. Ε, απλώς σε φάση σχεδιασμού είναι δυνατόν να σκεφτούμε και άλλους τρόπους εναλλακτικούς, όχι μόνο το αματέους αλλά και άλλα μέσα. Αυτή όμως είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία. Ε, βεβαίως πολλά μπορούμε να διδαχτούμε και όντω διδαχτήκαμε και προσπαθούμε να επιταχύνουμε με πολλά σχέδια και μέτρα μια καλύτερη διαχείριση των ορομοταφορών στην ε, Ευρώπη. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι τα ηφαίστεια δεν υπακούν ε, κανένα κανόνα ε, και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον τέτοια έκτακτα γεγονότα. Πάντοτε υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό είναι ένα ρίσκο που είναι μέρος του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Commissioner. Η συζήτηση έληξε εδώ. Η επόμενη συνεδρία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, 19 Μαΐου, από τις 9